afternoon, Καλό απόγευμα. Ε, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Ας ξεκινήσουμε τις εργασίες αυτής της ε, συνεδριάσεως. Έχουμε στην ημερήσια διάταξη ε, θέματα που είναι πολύ δεσμευτικά και που αναφέρονται εις ε, την παραγωγή ε, διοξίνη στο Τάραντο και έχουμε τον κύριο Ταγιάννη ε, εδώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπάρχει ένα θέμα για την, το κυνήγι της Φώκιας με τον Καναδά. Το θέμα ε, μία χωματερής στη Γαλλία, θέματα οικοδομικών επιχειρήσεων και νομοθεσίας στην Ισπανία. Ε, για τα ναυπηγεία της Μάλτας και για την ασφάλεια των ε, πυρηνικών ε, εργοστασίων και το τελευταίο αύριο είναι για την αξιοποίηση του αερίου από σχιστόλιθο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω αν έχει κανείς αντίρρηση και εφόσον δεν υπάρχει εγκρίνεται η μερίσια διάταξη με ορισμένες αλλαγές που αναφέρονται στο σημείο 7 το οποίο θα μεταφερθεί και θα αναβληθεί μέχρι την επόμενη συνεδρίαση λόγω ετήσεως της υπογράφου την αναφορά και το σημείο 9 το οποίο θα συζητηθεί πριν από το 8. Σας ενημερώνω ότι θα παραστούν οι, ε, αυτοί που έχουν προσυπογράψει τα σημεία 4, 6, 14, 15 και 19. Όπως σε κάθε συνεδρίαση ε, έχουμε διανύμει το παράρτημα εις ε, το έγγραφο της Προεδρίας και είδαμε ότι ε, δεν υπήρχαν σχόλια σχετικά με τα πρακτικά, οπότε θεωρούμε ότι υιοθετούνται. Κάποιος ζητάει το λόγο αυτή τη στιγμή. Βλέπω το σημείωμα της Προεδρού ότι ζητάτε να ξανανοίξει η, ε, ε, η αναφορά 1266 κάθετος 11 και πριν από δύο εβδομάδες είχαμε αποφασίσει να την κλείσουμε. Και ο μόνος λόγος να ξανα, ξανανοίξει μία αφορά, αναφορά είναι αν υπάρχουν ε, νέα στοιχεία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο νέο στοιχείο είναι η κατηγορία για δύο ευρωβουλευτές σχετικά με το θέμα αυτό. Αν όντως έτσι είναι, ε, ενίσταμε διότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται κάτι τέτοιο. Εάν ε, η κατηγορία είναι η μόνη αιτία της ε, να ξαναεξεταστεί αναφορά, δεν πρέπει να ξανανοίξει διότι δεν μπορούμε να υιοθετούμε τέτοιες πρακτικές. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ίσως καλό θα ήταν ε, να λάβω το λόγο αφού διακρίσει το θέμα που έθεσε ο κύριος Βαλές, αλλά αυτό το που με εξέπληξε εμένα προσωπικά είναι ότι υπάρχει αυτή η πρόταση να ξανανοίξει ένα θέμα που καταλαβαίνω ότι είχε κλείσει και έπρεπε να είχε κλείσει οριστικά μάλιστα. Για ποιο λόγο. Γιατί όπως είπε ο συνάδελφός μου δεν υπάρχει ούτε ένα επιχείρημα για να ξανανοίξει να διατηρηθεί. Εκτός από δύο επιχειρήματα τα οποία νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε, είναι και πάρα πολύ κακόβουστα θα έλεγα τα επιχειρήματα. Γιατί αναφέρθηκε και στην συνάδελφο Αγιούσο και σε μένα προσωπικά ο αναφέρον. Ε, για την κυρία Αγιούσο, ήδη από την πρώτη στιγμή πιστεύω ότι θα έπρεπε η αναφορά να είχε απορριφθεί, διότι ουσιαστικά αμφισβητεί την πάρα πολύ αναλυτική, αιτιολογημένη και επικυρωμένη και από νομική ε, γνωμάτευση ε, έκθεση της κυρίας ε, Αγιούσο για το ότι δεν υπάρχει ουδετερότητα ότι υπήρξαν κάποιοι που αποφελήθηκαν μόνο και μόνο γιατί ε, με τον ιδιοκτήτη του Europark που της πιάνει το χέρι εμφανίστε σε αυτό το γραφείο. Ποτέ στη ζωή δεν θα είχα φανταστεί ο κύριος Λόου για παράδειγμα ή η κυρία Κιώτη να μου πει ότι ξέρετε να στη σελίδα 4 ορίστε είστε σε μια φωτογραφία και παρά είστε φιλικοί όπως ε, ο κύριος ε, Κίσλιν πριν κυρία Αγίους, ακόμα πιο φιλικμά, ποτέ δεν θα είχα σκεφτεί ότι κάτι πιο πέρα συμβαίνει, ότι δεν είναι ευαίτερη, δεν είναι αμερόληπτη ή ότι θέλει να προωθήσει κάποιο φίλο. Είναι δυνατόν, δεν μπορούμε να δεχθούμε με τέτοια επιχειρήματα να ξανανοίξει αυτή η αναφορά. Επίσης θεωρώ απαράδεκτο και απίστευτο το γεγονός ότι εγώ που στην κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων το 97, 14 χρόνια, 15 χρόνια δηλαδή. Είχα ένα αξίωμα, ήμουν δηλαδή συμβουλο για θέματα γεωρία, στενοτροφίας και αλεία, να λέγεται ότι εγώ είχα θέση, σχέση με αυτό το πάρκο. Η μόνη σχέση που είχα με το πάρκο είναι αυτή που είχαν οι εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του πάρκου. Ακριβώς η ίδια σχέση. Ξέρω λοιπόν ότι Κανένα απολύτω συμφέρον δεν έχω με το πάρκο. Αυτοί σίγουρα έχουν κάποιο διαφορετικό συμφέρον. Και δίνει λοιπόν τρία επιχείρηματα αναφέρον. Λαμβάνεται μονομερή απόφαση χωρίς σε καμία περίπτωση να προασπίζονται τα συμφέροντα του ζώου. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας εδώ, κύριε Άουκεν, κύριος Μαρτίνεθ, κυρία Γιούσο, τα δικαιώματα των ζώων προασπίζονται. Το ίδιο κάνω και εγώ. δεν υπήρξε κάποιο άλλο εμπειρογνώμων σε θέματα φώκιας, λένε, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε αυτοί. Οι μόνοι δηλαδή εμπειρογνώμονε για θέματα φώκια είναι οι ίδιοι και δεν πήγαν. Δεν υπάρχει κανένα άλλο εμπειρογνώμων. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρα τα στοιχεία. Όλα τα επιχειρήματα έχουν τεθεί επιτάπητος και υπάρχει και απόφαση των ε, Ολλανδικών δικαστηρίων όπου επικυρώνονται όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποίησαμε για να λάβουμε τη σχετική απόφαση. Άρα, ειλικρινά δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση να τεθεί θέμα να ξανανοίξει αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ. Uh, Κύριε Άουκεν, εγώ θα έλεγα να το συζητήσουμε συνεδρίο των συντονιστών. Γιατί δεν μπορεί να ξεκινά τώρα μια πολιτική αντιπαράθεση και για διαφορετικές ε, απόψεις και γνώμες. Ε, αυτό είναι λίγο ονοχλητικό. Δεν μπορούν δύο μέλη να αποφασίζουν ότι όλα έχουν αποφασιστεί και έχουν γίνει. Νομίζω ότι αυτή η απόφαση πρέπει να ληφθεί στην συνεδρίαση των συντονιστών και εμεί να προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Η κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν ε, θέλω να προσθέσω τίποτα περισσότερο σε αυτά που μόλις προείπε ο κύριος Μάτου. Εγώ ήμουν παρούσα στην ε, παρουσίαση μιας ε, ταινίας για το περιβάλλον, ήταν εκεί και ο ιδιοκτήτης του πάρκου και τραβήξαμε μια, μια φωτογραφία οικογενειακή στο τέλος. Αν το επιχείρημα του κυρίου αυτού είναι ουσιαστικά ε, να προσπαθεί να δυσφημίσει για να μπορέσει να δικαιολογήσει αυτά τα οποία λέει. Δεν υπάρχει καμία βάση. Ούτε υπάρχει μία έκθεση, ούτε μία που να μην λέω ότι θα πρέπει να γυρίσει η φώκια στην θάλασσα. Όπως η όρκα που γύρισε για να πεθάνει στη θάλασσα και αυτό κόστησε 2 εκατομμύρια ευρώ. Η βιολογία της λόγω φάλαινας είναι περίπλοκη και έχω μάθει και εγώ πολλά και πολλοί κόσμος επίσης μπορεί να μάθει πολλά. Κύριε Στουργκάη, θα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν συμφωνώ με την κυρία Άου και να αποφασιστούν τα σχετικά στις συνεδρίες των συντονιστών. Εδώ πρέπει να κλείσει το ζήτημα. γιατί θα πάρει πολλές συνεδριάσεις συντονιστών για να αποφασίσουμε εκεί. Επίση, τα συζητήσαμε και κλείσαμε οριστικά το θέμα στην Επιτροπή μα. Νομίζω λοιπόν ότι ως τη Επιτροπή πρέπει να σα ζητήσω να κλείσετε ολοκληρωτικά πλέον την αναφορά αυτή. Και τι θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να μα ενημερώσει η γραμματέα τη Επιτροπής μα για ποιο λόγο ελήφθη η απόφαση να ξανανοίξει η αναφορά αφού, όπως είπατε, πραγματικά ε, έχουμε όλες αυτές τις ε, εξελίξεις. Έρχεται εκ των υστέρων αναφέρον, δηλαδή, που δεν του αρέσει η απόφαση που λάβαμε εδώ και η ψηφοφορία δεν του αρέσει και μας ζητά να ξανανοίξουμε την αναφορά ή οποιαδήποτε άλλη αναφορά. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Νομίζω ότι κυρίαρχη είναι η Επιτροπή μας για να λαμβάνει αποφάσεις. Έλαβε λοιπόν απόφαση για αυτό το θέμα. Τελεία και παύλα. Ο κύριος Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι η γραμματεία αυτό που έκανε ήταν ότι από τη στιγμή που υπήρξε αίτηση του αναφέροντος, φυσικά και η γραμματεία δεν λαμβάνει απόφαση να ξανανοίξει η αναφορά, απλά θέτει αυτό το ζήτημα, όπως οφείλει. Εδώ και όχι στους συντονιστές, θέτει αυτό το θέμα. Θα ανοίξει ή δεν θα ξανανοίξει η αναφορά. Ακούστηκαν οι απόψεις πολλών από εμάς που είπαμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι σκόπο να ξανανοίξει αναφορά. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε, και είναι ένα θέμα κυρία Πρόεδρε που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αν η γραμματεία πρέπει να έχει, αν θέλετε, τη νομική ε, δυνατότητα και εξουσία να απορρίπτει την αναφορά ενός αναφέροντος, όπως στην προκειμένη περίπτωση, Μία αναφορά ενώ που δεν δίνει κανένα καινούριο στοιχείο, καμία καινούρια πληροφορία σε μία υπόθεση που την αναλύσαμε και την ξανααναλύσαμε, αυτό νομίζω ότι ε, αποτελεί προσβολή. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο εκφράζει το αναφέρον είναι προσβολή. Δεν μπορεί. Επειδή κάποιος έχει ή είχε κάποια στιγμή ασκήσει ένα αξίωμα να τον κατηγορούμε ακούσαμε, αναλύσαμε, ακούσαμε πυρογνώμονες. Εγώ δεν είμαι πυρογνώμων, σέβομαι πάρα πολύ τους κυρίους ε, Μάτο Βαλέση και την κυρία Γιούσο και τις ε, γνώσεις τους. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα επιχείρημα και να κατονομάζεται κάποιος να λέει ο τάδε κύριος που ήταν σύμβουλος πριν από 15 χρόνια, ε, γιατί είναι ακόμη σύμβουλος. Μα όλα τα είδαμε πάρα πολύ σοβαρά, σε πολύ μεγάλο βάθος και με πολύ μεγάλη προσοχή. Ίσως η γραμματεία θα μπορούσε να έχει απαντήσει λέγοντας ότι λόγω των επιχειρημάτων ακριβώς ούτε καν θα τεθεί ζήτημα να ξανανοίξει αναφορά αυτή. Η γραμματεία είπε ότι η, Ευρωπαϊκή, η, Επιτροπή μας είναι αυτή που θα αποφασίσει, έτσι έκρινε και νομίζω ότι πράγματι πρέπει τώρα να αποφασίσουμε να μην ξανανοίξουμε την αναφορά αυτή. Είναι ένα θέμα, επαναλαμβάνω, που συζητήθηκε ξεκάθαρα και φαίνεται ότι οι παρόντες τουλάχιστον στην πλειοψηφία μας, γιατί εμείς αποφασίζουμε, θεωρούμε ότι το ζήτημα έχει λήξει, έχει κλείσει αναφορά. Και πρέπει να απαντήσουμε στον αναφέροντα ότι η Επιτροπή μας, αφού μελέτησε και τα δικά του στοιχεία, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να τα κρίνει παραδεκτά αυτά τα επιχειρήματα. Επομένως, έχει κλείσει το ζήτημα. Εντάξει, ίσως υπάρχει μια ψήφος κατά. Θα δούμε. Ευχαριστώ κύριε Μαρτίνες. Ορίστε, κύριε Άοκεν. Τώρα συζητάμε το θέμα πραγματικά και τα μόνα επιχειρήματα τους είναι αυτά. Δεν προσπαθώ να προσβάλλω κάποιον. Θέλω να πω ότι δεν ακούσαμε κάποιον ειδικό απ' έξω. Και ενώ μεταξύ εγώ αυτό έκανα. Ξέχασα το αγγλικό όνομα του ζώου, του κήτους, αλλά αν είναι τόσο νέα, είναι κανονικό να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Αυτό κάνουν. Και έχουμε πολύ καλούς εμπειρογνώμονες στη Δανία. Αιώνες ασχολούμαθα με τη φαλαινοθυρία και ξέρουμε πολλά. Μόνο η ισπανική υπόθεση. Αν μια χώρα αισθάνεται ότι έχει τους δικούς της εμπειρογνώμονες και είναι προσβλητικό ότι ζητάμε άλλους εμπειρογνώμονες, πέραν των δικών τους, τι να πω, αν αυτή η θέση είναι θέση κατά της οποίας διαμαρτύρομαι και αισθάνομαι ότι καταστρέφεται, καταστρέφεται το έργο της Επιτροπής μας. Διότι αυτή η ειδική δεν είναι η μόνη ειδική στον κόσμο και έχουμε και αμερόληπτους εμπειρογνώμονες εκτός Ισπανίας. Υπάρχουν. Ευχαριστώ, κυρία Όκεν. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τη θέση της πλειοψηφία της Επιτροπής. Θα ήθελα να διευκρινίσω αυτό που έθιξε ο συνάδελφος Μαρτίνες, κάτι που εμπεριέχεται και στα όσα είπαν οι άλλοι συνάδελφοι. Δεν αποφασίζει η γραμματεία, υπάρχει μια διαδικασία που εφαρμόζουμε στην πράξη όσον αφορά νέα έγγραφα που καταφθάνουν στην Επιτροπή Αναφορών και η Γραμματεία κάνει μια πρόταση. Η πρόταση διανεμήθη στα μέλη της Επιτροπής, τα οποία έχουν το χρόνο να εξετάσουν τα κείμενα και να αποφασίσουν. Εν τη αυτή περιπτώση, είμαστε στην ώρα των ψηφοφοριών. Ε, εκφράστηκαν όλοι εκτός από την κυρία Άοκεν, Όλοι οι άλλοι υπέρ του να μην ξανανοίξει αυτή η αναφορά, θεωρώντας ότι το αντικείμενο των νέων πληροφοριών επί των οποίων θα βασιζόταν το άνοιγμα είναι απλώς μια ανακοίνωση γνωστού της κυρίας Αγιούσο με το κίνημα που ενδιαφέρεται αυτό το θέμα. Δεν είναι επί της ουσίας κάτι καινούριο που επιτρέπει να ξανανοίξει η αναφορά. Οπότε αποφασίζουμε με την πλειοψηφία των παρόντων αυτή η αναφορά να μην ξανανοίξει. Δεν είχαμε άλλε αντιρρήσει για τα υπόλοιπα. Δεν βλέπω συναδέλφου να ζητούν το λόγο. Η πρόταση περιέχεται στο προσαρτημένο φάκελο με το έγγραφο του Προέδρου. Θεωρείται ότι εγκρίνεται. Διανεμήθη μετά και ο κατάλογος των ούτως αποκολωμένων ετοιμάτων ε, συζητησίμων ε, και εδώ υπάρχει η πρόταση που ετοίμασε η γραμματεία. Εκεί χρειάζεται η γνωμοδότηση των μέλων της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να εκφράσουν την άποψή τους μέχρι τις 18, στις, μέχρι Τετάρτη 10, 6 ώρα το απόγευμα. Αν δεν παρέμβουν οι συνάδελφοι, η πρόταση θα θεωρηθεί εγκεκριμένη ως διανεμήθη στα μέλη της Επιτροπής. Όσον αφορά τις ανακοινώσεις, το σημείο 3 να σας πω ότι θα χάσω άλλο μέλος της γραμματείας διότι θα μεταφερθεί σε πιο καλή θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κάρολιν Λέφλερ ήταν μαζί μας για πάνω από τρία χρόνια και θα αναλάβει καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι θα συμφωνούν ότι πρέπει να την ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που έκανε σε αυτή την Επίτροπη και πάνω απ' όλα της ευχόμαστε καλή δουλειά στην επόμενη θέση της ε, και σε ευχόμαστε το καλύτερο για το μέλλον της. Στις 17, στις 5 θα διακοπούν οι εργασίες της Επιτροπής για να ξεκινήσουν οι εργασίες των συντονιστών, η μερίσια διάταξη των συντονιστών είναι στο φάκελό σας που διαναμήθη. Αυτές τις πληροφορίες σας τις δίνω, διότι το πρώτο σημείο της συνεδριάς των συντονιστών είναι η παρουσίαση της διαδικασίας όσον αφορά την πύλη την, στο διαδίκτυο της Επιτροπής που μπορεί να ενδιαφέρει και άλλους συναδέλφους. Οπότε για αυτό το πρώτο σημείο καλείστε αν θέλετε συμμετάσχετε στις συνεδρία των συντονιστών. δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις. Οπότε πάω στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, την πρώτη αναφορά της ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη αναφορά είναι η 1044 του 2011 που υπευλήθη από τον Ζωάννα Σβάμπερ, Βρετανίδα οικοών, ε, ονόματι μιας οργανώσεως που είναι the Human Society International. Η αναφορά ε, υποστηρίζεται από άλλους 22 και το αίτημα να δημιουργηθεί ένα Συμβούλιο Διαμεσολάβησης του ΠΟΕ βάσει του 1007 του 2009 και του Συμβουλίου της 16 Σεπτεμβρίου του 2009 όσον αφορά το εμπόριο από προϊόντα φώκιας. Θέλω να συζητηθεί κατά πόσο εφαρμόζεται σωστά ο λόγο κανονισμός. Είναι παρούσα ε, η αναφέρουσα, οπότε της δίνω το λόγο για ένα πεντάλεπτο. Η Τζοάννα Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Humane Society International και πάνω από 20.000 ανθρώπους που έχουν υπογράψει, πέρα από τους 22 όταν υποβάλαμε την αναφορά, θέλω να σε ευχαριστήσω κυρία Ματσόνη για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε στην Επιτροπή για δεύτερη φορά για το συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά την αναφορά μας για την πρόκληση κατά, που αμφισβητεί ο Καναδάς τον κανονισμό όσον αφορά ε, το εμπόριο προϊόντων φώκες στον ΠΟΕ. Ε, είναι επίκαιρο ότι είμαι εδώ στα μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Πριν από δύο εβδομάδες οι καναδικές, η καναδική και νορβηγική κυβέρνηση ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν με την προσφυγή του στον ΠΟΕ και θέλουν γρήγορα να δημιουργηθεί ένα πάντα στον ΠΟΕ για το θέμα αυτό. Εξακολουθούν να διατείνονται ότι αυτή η νομοθεσία δεν ταιριάζει με τους κανόνες του ΠΟΕ και το εμπόριο των ε, προϊόντων φώκιας θα πρέπει να αποκατασταθεί. Υιοθέτησε την απαγόρευση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά η παγκόσμια αγορά για τα, τα προϊόντα της εμπορικής φαγής των, ε, της φώκιας απαγορεύθηκε και απαγόρευσε την εισαγωγή ε, από γούνες η Ρωσία. Ε, οπότε έκλεισε και άλλη μια σημαντική αγορά και η Ταϊβάν επίσης εισάγει μια απαγόρευση όσον αφορά το εμπόριο ε, των προϊόντων αυτών και τον επόμενο μήνα ακόμα και η, Σουηδική, η ερβετική ε, Γερουσία ε, θα εισάγει απαγόρευση γιατί το Κοινοβούλιο θέλει να απαγορεύσει τα απάνθρωπα αυτά προϊόντα που προέρχονται από το εμπόριο φώκιας. Το εμπόριο προϊόντων φώκιας πεθαίνει τόσο πολύ που φέτος η καναδική κυβέρνηση έδωσε 3,6 εκατομμύρια δολάρια στον τομέα της φώκιας για να παραμείνει ε, ζωντανή και στον τομέα μεταποίησης ε, δέρματο ε, φώκια. Παρόλο που έμεναν απούλητες γούνε και δέρματα από την περσινή χρονιά του κυνηγίου. Παρόλα αυτά, το τρόπο που σφάζονται οι φώκες δεν είναι πιο ανθρωπιστικός, δεν ρυθμίζεται καλύτερα από όταν είχε αποφασίσει το Κοινοβούλιο να, αποφασ... να απαγορευτούν το 2009 τα πρώτα τη φώκιας. Το βλέπουμε και στι ταινίε που δείχτηκαν πρόσφατα. Εξακολουθούμε να έχουμε στοιχεία ε, των διαφόρων των μικρών της φώκιας που τα καμακώνουν και τραβάνε πάνω στον πάγο ή τα ανεβάζουν πάνω στα πλοία ενώ ψυχοραγούν. Και βλέπεις τα μικρά που ψυχοραγούν και φωνάζουν πάνω, σορευμένα πάνω στα πτώματα των άλλων ζώων. Ε, και φώκες πυροβολούνται και μένουν στην αγωνία, την επιθανάτια. Και βλέπουμε ε, στο νυχτό, στην ανοιχτή θάλασσα να πυροβολούνται επανειλημμένα οι φώκες. Είναι πολύ αποκαδιωτικές αυτές οι εικόνες θα συμφωνείτε. Λόγω όμω του κλεισίματο τη αγορά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, πολλέ χιλιάδε φώκε σώθηκαν από αυτή την κακή μοίρα. Αλλά συνεχίζεται αυτή η απάνθρωπη μεταχείριση, όμω η κλίμακα ε, βασάνων των ζώων έχουν, έχει μειωθεί λόγω αυτών των μέτρων. Είμαστε τα μάλα απογοητευμένοι που ο Καναδάς εξακολουθεί να προσφεύγει κατά του κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για τα προϊόντα φώκια στον ΠΟΕ. Θεωρούμε ότι αυτή η προσφυγή στον ΠΟΕ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια άμεση επίθεση κατά των ηθικών αξιών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά των ευρωπαϊκών δημοκρατικών μας διαδικασιών. Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι η νομική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπερασπίστηκαν στεναρά τον κανονισμό, ή μάθε υπερασπιστούν στεναρά τον κανονισμό όταν θα εξεταστεί το θέμα στον ΠΟΕ. Όμως, αυτό που εμείς σαν πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως θέλουμε και ανησυχούμε γι' αυτό, είναι ότι θέλουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βλέπουμε ότι διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Καναδική κυβέρνηση χωρίς να θέτει όρο την απόσυρση του Καναδά από την έφεση που έχει, την προσφυγή που έχει κάνει στον ΠΟΕ. Αυτό κατά την άποψή μα είναι απαράδεκτο να συναυθεί τέτοια συμφωνία εμπορική ενώ ταυτόχρονα ο Καναδά ε, κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να καθορίζει δημοκρατικά ποια προϊόντα επιλέγει να εμπορεύεται βάσει των δικών μα ηθικών ευαισθησιών. Τελευταία φορά που μίλησα στην Επιτροπή σα, ο εκπρόσωπο τη γενική Διευθύνσεως ε, Εμπορίου είχε, ο είχε εξοργιστεί. Και έλεγε ότι η προσφυγή του ε, Καναδά στον ΠΟΕ ήταν κάτι εντελώ ξεχωριστό από τι διαπραγματεύσει εμπορικέ. Το θέμα είναι ότι αν εσεί, σαν ευρωβουλευτέ, το ίδιο αισθάνεστε, αυτή είναι η άποψή σα. Ε, πέρσι, το Κοινοβούλιο εθέτησε ένα ψήφισμα για τι εμπορικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά και εκεί αναφερόταν ότι η προσφυγή στον ΠΟΕ αντιβαίνει των θετικών εμπορικών σχέσεων και θέτει την κατακύρωση, υπονομεύει την ε, επικύρωση συμφωνία ΣΕΤΑ. Και πάνω από 100 ευρωβουλευτέ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προ την καναδική κυβέρνηση που εξέφραζαν το ότι προτίθεται να καταψηφίσουν τη συμφωνία ΣΕΤΑ λόγω του θέματο τη φώκιας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε επίσημα να διαχωρίσει τα δύο θέματα, παρά την απογοήτευση ευρωβουλευτών, που κάποιοι από αυτούς πιστεύω ότι είναι παρόντες. Όμως, πέρα από τις φώκες, Επίση, υπάρχουν και απαιτήσει για θεωρήσει διαβατηρίων των Τσέχων και των Βουλγάρων υπηκών που να στον Καναδά. Και αυτό υπονομεύει την εμπορική συμφωνία. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το προσέξουμε. Ε, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλά διακυβεύονται εδώ, περισσότερα πέρα από την απαγόρευση των φώκια από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά πολύ και την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου στα μάτια των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το Κοινοβούλιο δεν υπερασπιστεί την ομοθεσία του, οι απλοί πολίτε σίγουρα θα χάσουν κάθε εμπιστοσύνη στην πολιτική διαδικασία. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να μου πει πώ εμεί, αν πολίτες Μπορούμε να εμπιστευόμαστε το Κοινοβούλιο εάν δεν καταφέρνει να προσπιστεί στεναρά νομοθεσία για την οποία είναι υπεύθυνο και ανταυτού συμφωνεί χωρίς αμφισβητήσεις επί συμφωνίας να δώσει δισεκατομμύρια σε μια χώρα που δεν σέβεται τι ηθικέ μα αξίε. Με την επικύρωση τη συνθήκη Αβώνα, το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να δείξει ότι είναι ισχυρό και να επιβάλλει τη θέλησή του. Ε, θα θέλαμε, από εσά εξαρτάται να το κάνετε αυτό. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ έντονα με αυτά τα οποία είπε η αναφέρουσα. Είναι ξεκάθαρε οι απόψει μου για ε, τον τρόπο με τον οποίο θανατώνονται οι φώκε. Έχω δει να τις ε, δέρνουν ζωντανές. Και πραγματικά το βάσανό τους δεν παίρνει ε, τέλος. Ώρες κάνουν για να σοφήσουν. Το κοινοβούλιο έχει εγκρίνει μια γραπτή δήλωση για τη θανάτωση φώκιας Είμαστε αντίθετοι λοιπόν ε, στη θανάτωση της ε, φτώχεια και στους Καναδούς. Πολύ ξεκάθαρο όπως υπόθηκε σε πρόσφατη δήλωσή μας. Είπαμε ότι θα θέσουμε που αυτή την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τον Καναδά, ΣΥΤΑ, εάν συνεχίσουν τη διαδικασία προσφυγής στον ΠΟΕ. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προασπίζεται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε νομοθέτημα στο διεθνέ προσκήνιο θα πρέπει να το υποστηρίζουμε. Το συγκεκριμένο όμω νομοθέτημα είναι ένα θέμα ε, πολύ λεπτό για το Ευρωπαϊκό κοινοβόλιο, πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα και πρέπει να ασκήσουμε πίεση. Έχουμε διπλό καθήκον να προστατεύσουμε αυτό το νομοθέτημα και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στου καναδού ότι δεν ε, μας αρέσει καθόλου η διαφορά αυτή ε, στο επίπεδο του ΠΟΕ. και πρέπει να πούμε ότι ε, αυτό το οποίο ισχυρίζονται ότι δεν έχει καμία σχέση αυτή η προσφυγή με την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, εμάς μας βρίσκει αντίθετος, εμείς θεωρούμε ότι είναι συνδεδεμένα άρρηκτα αυτά τα δύο. Πρόεδρος. Συγγνώμη, αλλά υπήρξε ε, μια... Δεν, δεν, κατάλαβα καλά με τον κύριο Λό ακριβώς τι έγινε. Πρώτα έπρεπε να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της ε, Επιτροπής, ο Κόλλιν Μπράουν, λοιπόν, ε, θα λάβει πρώτο το λόγο και μετά οι υπόλοιποι βουλευτές. Κύριε Μπράουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε σε αυτή την Επιτροπή και να αναφερθούμε στις ανησυχίες που εξεφράστησαν στην αναφορά. Ήθελα να αναφέρω τέσσερα σημεία, ακροφυγώς, πρώτα απ' όλα. Όπως είπε η κυρία Σουάμπ, επιβεβαιώνω ότι ο Καναδάς πράγματι ξαναπρόθεσε την υπόθεση στον ΠΟΕ μαζί με την Ορβηγία. Σημαντικό θέμα αυτό. Έχουν ξαναθέσει το ζήτημα τις τελευταίες 15 μέρες. Τα τέσσερα σημεία που ήθελα να θίξω ακροθυγός. Λοιπόν, πράγματι, και το επαναλαμβάνω αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως θα προασπιστεί στεναρά αυτή την νομοθεσία, όπως πολλά από τα μέλη σας γνωρίζουν, είχαμε εμπλακεί μέσω της υποβολής της προτάσεως, αλλά θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι η υιοθετηθήσα νομοθεσία συνάδει με τον ΠΟΕ. Και έχουμε την πεποίθηση ότι θα επιβιώσει έναντι ασδήποτε προκλήσεως. Δεύτερον, πράγματι, και σκαταγραφεί στα πρακτικά, Τίποτα στην Συμφωνία Ελευθερεμπορίου με τον Καναδά δεν θα υπονομεύει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να διατηρήσει αυτό το νομοθέτημα. Τρίτον, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρούμε ότι είναι καλό να επιδιώξουμε διαπραγμάτευση αυτής της διαφοράς στα πλαίσια της εμπορικής συμφωνίας. Αυτό θα ειδωθεί κατά την άποψή μας από τον Καναδά σαν ε, δείγμα δυναμίας. Και να υπενθυμίσουμε ότι βεβαίω η νομοθεσία για τις φώκες είναι πολύ σημαντική, όμως έχουμε άλλες προσφυγές κατά του Καναδά που έχουμε κάνει εμείς και που εξετάζονται από το σύστημα του ΠΟΕΤ και τώρα που μιλάμε. Και ενώ διαπραγματευόμαστε την προναφερθήσα συμφωνία. Τέταρτον, να υπενθυμίσω, όπως ανέφερε και αναφέρουσα, ότι δεν είναι μόνο ο Καναδάς που έχει προσφύγει αλλά και η Νορβηγία. Άρα πρέπει να μας προβληματίσει το πώς, πώς θα μπορέσουμε να χωρίσουμε τον Καναδά και την Νορβηγία. Ο μόνος τρόπος για να τους χωρίσουμε είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει όσον αφορά την νομοθεσία για τις φώκες. Αυτό θέλουν, είναι απαράδεκτο αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν βλέπουμε καμία προοπτική να βρούμε ενδεχόμενη λογική λύση που θα λαμβάνει υπόψη και τον Καναδά και την Ορβηγία. Τέλος, να πω ότι βεβαίως ε, σημειώνουμε την έκκληση που απίθυνε στο Κοινοβούλιο για να φέρουσα να υπερασπιστούμε την ομοθεσία μας και γνωρίζουμε πολύ καλά όπως είπε ο κ. Μάρτιν, ποιος είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου όσον αφορά αυτή την νομοθεσία. Η νομοθεσία εγκρίθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, νομοθέτημα του Κοινοβουλίου, αλλά και εν μέρη και νομοθέτημα του Συμβουλίου. Και έχει επιφορτιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εφαρμογή της νομοθεσίας και η προάσπισή της είναι κάτι που έχει τεθεί και σε επίπεδο εξωτερικών σχέσεων. Σας διαβεβαιώνω, διαβεβαιώνω την Επιτροπή σας, θα υπερασπιστούμε στεναρά, γενναία αυτή τη νομοθεσία στη διαμάχη με τον Καναδά, που δυστυχώς αποφάσισε να προχωρήσει με αυτή την προσφυγία. Ευχαριστώ. κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Και ε, ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο δόκτωρα Σουέιπ και οι, συνάδελφοι. Διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Κοινοβούλιο συναισθάνεται πολύ σημαντικά το θέμα αυτό. Από το 1983 έχουμε ε, προβεί στην ψήφιση ε, οδηγιών εναντίον αυτών των εισαγωγών και το 2008 παραδείγματος χάρη ε, η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απαγορεύσει την εισαγωγή προϊόντων φώκιας και ζήτησε να υπάρξει μία ισχυρή απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων φώκιας. Άρα η αντίθεση είναι προφανές. Το Κοινοβούλιο έχει αποφανθεί. Βλέπω ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αναφορά λέγει ότι δεν μπορούν να συνδεθούν τα δύο θέματα. Δηλαδή δεν μπορούν να ζητήσουν από τον Καναδά να αποσύρει ε, την ε, προσφυγή στον ΠΟΕ. Και πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα δεν θα εξαλειφθεί και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πιστεύει ότι θα μπορέσει να νικήσει και ότι θα μπορέσει να πείσει τους Καναδούς να αποσύρουν το αίτημα. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αλλάξει η αντιμετώπιση και αντί να ζητήσει από τους Καναδούς να αποσύρουν την ε, προσφυγή στον ΠΟΕ, να ζητήσει να μην κυρώσει την ε, ΣΥΤΑ μέχρι ότου η ενέργεια αυτή να έχει επιληθεί στον ΠΟΕ. Γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρόκειται ε, για μια επιχείρηση και ε, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι στέλνουν θαλάσσιες ε, ε, ζωοτροφές και θαλάσσια είδη τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα χαθούν 6 εκατομμύρια ευρώ εξαγωγών ετησίως. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί να αποδείξει πόσο σημαντική είναι αυτή η νομοθεσία όσον αφορά την αλία. Και επιπλέον, εάν μπορούμε να επηρεάσουμε τους Καναδούς και να μην κυρώσουν τη ΣΥΤΑ μέχρι ότου λυθεί το θέμα του ΠΟΕ, ενδεχομένως θα κερδίσουμε και το Κοινοβούλιο θα επιτύχει αυτό που επιζητεί από το 1983. Θα παρακαλούσα λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά για να εξετάσουμε την ιδέα αυτή και να προσπαθήσουμε να την προχωρήσουμε. Και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας κύριε με ενδεχομένως και γραπτός άμα θέλετε. Κύριος ματίνες Ματίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η αναφέρουσα παρουσίασε εξαιρετικά την αναφορά της με πολύ πιστικό τρόπο και αν χρειαζόταν κάτι αρκεί που είδαμε αυτή την ε, παρουσίαση με τις διαφάνειες που συμπλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα λόγια της αναφέρουσας με εντυπωσιακό τρόπο θα έλεγα. Κάθε φορά που βλέπουμε αυτό το θέαμα είναι αδύνατον να πιστέψει κανείς ότι μια χώρα όπως ο Καναδάς που μας φαίνεται ότι είναι άνθρωποι Καναδοί που σέβονται αρχές και μάλιστα πολλές φορές δίνουν και μαθήματα προς άλλες χώρες. Όταν όμως βλέπουμε στην πραγματικότητα τι καταγγέλλεται, είναι πραγματικά να σου σηκώνεται η τρίχα. Εξήγησε ο κύριος Μάρτιν ποια είναι η θέση μας για το θέμα αυτό και η πρόταση του κύριου Τέιλορ κατ' πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και σοβαρά μάλιστα. Πάντως, κυρία Πρόεδρε, για ένα τέτοιο θέμα, το οποίο έχει αποφανθεί πολλές φορές στο Κοινοβούλιο και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, δεν μπορεί να θεωρηθεί έλασον ζήτημα ή να ξεχαστεί γιατί δεν αφορά εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Είναι αρκετά σοβαρό από μόνο το αυτό το ζήτημα για να του δώσουμε προτεραιότητα και να το αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Όσοι είμαστε εδώ παρόντες σήμερα, νομίζω ότι για μια ακόμη φορά είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να δοθεί δίκαιο και να δικαιωθούν οι προσπάθειες της αναφέρουσας και όλων όσων αγωνίζονται μαζί της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως αφενός είναι μια λυπηρή κατάσταση διότι η διαδικασία αυτή μας ακολουθεί εδώ και χρόνια και αν δεν υπήρχε αυτή η απαγόρευση ε, τότε ε, θα είχε καταρρεύσει η αγορά για τα προϊόντα αυτά εδώ και χρόνια. Ε, οι Καναδοί μας λένε «Μα τι επιζητείτε, θέλετε ε, να σταματήσετε κάτι για το οποίο δεν υπάρχει πλέον αγορά». Τώρα υπάρχει και η απαγόρευση πέραν των άλλων και υπάρχει μία γνωμοδότηση και άλλης επιτροπής και ε, της Ολομελίας του Κοινοβουλίου οπότε τι πρέπει να γίνει καταρχήν να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εκεί που εγώ ε, ε, διαφωνώ, μάλλον να το πω διαφορετικά, ελπίζω ότι στο τέλος αυτής της διεργασίας θα υπάρξει μία συμφωνία για ελεύθερο εμπόριο και απαγόρευση για εμπορία αυτών των προϊόντων. Τώρα πώς αυτό θα επιτευχθεί έξυπνα και στρατηγικά ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αφήσουμε στη διάκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς θα κάνει τις προκατακτικές διαπραγματεύσεις της σας. Δηλαδή αν ε, θα πει στους ε, Καναδούς αποσύρτε την πρόταση του ΠΟΕ από τον και μετά θα μιλήσουμε μαζί σας. Και πρέπει να ενημερώσουμε και τις αρμόδιες επιτροπές που είναι ε, ουσιαστικά πιο ενήμερες για τα θέματα των Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία γρήγορη ενημέρωση ε, σε περίπτωση που στις διαπραγματεύσεις αυτές κάτι στραβώσει. Δεν θα ήθελα να υπάρξει μία Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και μετά να ξαναξεκινήσει η διακίνηση αυτών των προϊόντων στην Ευρώπη. Παρακαλώ λοιπόν ενημερώστε την αρμόδια επιτροπή, αφήστε ανοιχτή την αναφορά και αφήστε την ε, επιτροπή να δράσει ε, υποστηρίζοντας την όμως. Λοιπόν, ε, υπάρχει απάντηση από την αναφέρουσα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ευρωβουλευτές στήριξαν την αναφορά αυτή και να σας πω ότι σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Γιάννη έχουν ε, ε, μεταφραστεί σωστά για την στήριξη της ε, απαγόρευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εποχή εκείνη υπήρχε μια αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προωθεί το πολύ από τους κανόνες Καναδούς. Υπήρχε λοιπόν ένας λόγος για να δράσουμε. Δεν ήταν αμεληταία ε, η ποσότητα του εμπορίου αυτού και παρακαλώ όντως να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι υπάρχει πλειοψηφία στην Επιτροπή αυτή για να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά λαμβάνοντας υπόψη τις ε, ε, την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, Νομίζω ότι δεν υπήρξαν αντιρρήσεις, οπότε μπορούμε να προβούμε σε αποστολή ενός γραπτού σημειώματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να μην συναυθεί μία εμπορική συμφωνία, που ο Καναδάς να σεβαστεί την κοινοτική νομοθεσία. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις μπορούμε να στείλουμε το σημείωμα αυτό εις ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ την ε, εκπρόσωπο, ε, την υπογράφησα την αναφορά και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η 359 του 2011 της Κριστίνας Βέζικα με 870 υπογραφές η οποία αναφέρεται στην ε, ε, μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντολογική νομοθεσία της ε, πολωνικής πλευράς στην κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοαερίου. Είναι μία αναφορά στην οποία έχει γίνει μία πρώτη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν επισυναφθεί και διάφορα έγγραφα και σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά το Μάρτιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε μία γνωμοδότηση στην Επιτροπή μας λέγοντας ότι ναι, τα γεγονότα τα οποία καταγγέλλονται ε, δεν συνάδουν με τον κίνδυνο το οποίος ε, επισύεται. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν ε, άλλοι προσυπογράφοντες και δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενδεχόμενα σχόλια για να μπορέσουμε να πάρουμε μία απόφαση. κυρία Αλήσια Κοσλόφσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα υπέβαλε την απόφαση του Πολωνικού Δικαστηρίου που αποφάσισε να ακυρώσει την απόφαση της τοπικής αυτοδίκησης να μην, να μην απαιτείται μία απόφαση για επεξεργασία διαφόρων προτάσεων. Δεν έχει λήξει η, νομοθετική... η δικαστική διαδικασία στην Πολωνία η απόφαση του δικαστηρίου θα επέτρεπε στην αναφέρουσα να προχωρήσει περισσότερο στα εθνικά δικαστήρια. Στη συγκεκριμένη υπόθεση το Εθνικό Δικαστήριο ενετόπισε διαδικαστικές ανομαλίες όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών συνεπειών. Η οδηγία δυστυχώς δεν ξεκαθαρίζει τι πρέπει να συμβεί όταν κάτι τέτοιο προκύψει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεώρησε ότι η αξιολόγηση συνεπειών είναι μια διαδικασία που καταρχήν θα πρέπει να γίνει πριν να κατασκευαστεί ένα έργο και αυτό αντικατοφτρίζει τον, τον προληπτικό χαρακτήρα της οδηγίας. Όμως, όπως συγκεκριμένη περίπτωση, σε κάποιες περιπτώσεις, για κάποιο λόγο, μπορεί να γίνει ένα διαδικαστικό λάθος και η απόφαση του δικαστηρίου ε, λαμβάνεται αφού έχει ήδη οικοδομηθεί ένα έργο, κατασκευαστεί κάτι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν αναφέρει λεπτομερώς τι συμβαίνει αντί αυτή η περίπτωση. Αναγνώρισε όμως το δικαστήριο ότι οι εθνικές αρχές θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα σε εξαιρετικέ περιπτώσεις να διευθετούν τα ζητήματα. Σε αυτή την περίπτωση υποθέτουμε ότι η εκδικαζόμενη υπόθεση δεν έχει ε, ολοκληρωθεί, δεν έχει διεκπαιρεωθεί, άρα δεν είναι χρήσιμο να παρέμβει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πιθανότατα οι πολωνικές αρχές θα μας απαντήσουν να μην προσφύγουμε ότι συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία και ότι πρέπει να περιμένουν για το τελικό αποτέλεσμα, για το πόρισμα, για την απόφαση ε, των δικαστηρίων των εθνικών. Ευχαριστώ. Άλλος που θέλει να μιλήσει. Νομίζω ότι εν αναμονή της λήξης των διαφόρων διαδικασιών στις οποίες αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν καλό να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και μετά να κλείσει με αιτιολογημένα στοιχεία όταν θα έχουμε και άλλες πληροφορίες που θα μας έχουν χορηγηθεί Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση. Σας ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη αναφορά. Η κυρία Άουκεν. Πριν κλείσουμε το θέμα. Και πάλι είναι μια περίπτωση που δεν έχουμε δει τι θα γίνει με την Είπαμε να μην την κλείσουμε. Α, ναι, αφού πήραμε τα πώς να μην κλείσουμε, εντάξει, ωραία. Passiamo, passiamo alla petizione 751-2001. Πάμε στην 751-2011, το Jean-Louis Postet, γαλλική ηθαγένεια εξ ονομασίας της MOV Vivante. Υπάρχουν και άλλες δύο υπογραφές που συνοδεύουν την αναφορά και είναι σχετικά με την εικαζόμενη οδηγία οδηγίας 1999-31 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την υγειονομική ταφή αποβλήτων. Είναι παρόν λοιπόν ο αναφέρον, ε, στον οποίο δίνω το λόγο για ένα πεντάλεπτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές, κυρίες και κυρίους, να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταθέσαμε στις 22 Ιουνίου του 2011 αυτή την αναφορά και επιμείναμε στο ότι δεν τηρείται η οδηγία για τις ε, από τον ε, νομάρχη του περιοχής Λουάρη και από το γαλλικό κράτος, ιδίως ό,τι αφορά την ε, συγκεκριμένη χωροταφής ε, αποβλήτων που δεν σέβεται την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Συγκεκριμένα, ο υδροφόρος αυτός ορίζοντας, Μπός, πολύ γνωστός, μεγαλύτερος υδροφόρος, μεγαλύτερη δεξαμενή υδατός στη Γαλλία που πρέπει να προστατευτεί και επειδή υπάρχει ε, το δάσος ε, Σεν Λιφάρ, το βλέπετε στο χάρτη αυτό. Είναι ένα χώρο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, λόγω της χλωρίδας και της πανίδας. Και βλέπετε εκεί αριστερά την εθνική οδό που πηγαίνει από την Ολεάν στη Μάγνου. Και είναι μέσα στην προστατευόμενη αυτή περιοχή. Ακριβώς επίσης λόγω του ότι αυτή, αυτή, αυτή η σοχήτα είναι κοντά ε, σε προστατευόμενα είδατε γιατί εκβάλλουν στον ε, Λίγυρα. Έχουμε στη διάθεσή σας στοιχεία, έχουμε αυτό το έγγραφο που έγινε το 2011 ε, και δείχνει ότι υπάρχουν οικοσυστήματα, βιότοποι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη ζώνη παρέμβαση. Είμαστε δύο ενώσεις, ε, Βιβάντ, Vivant, πρόεδρος της οποίας είμαι εγώ και περιλαμβάνεται στο France Nature Environnement και είναι και η Ένωση των Φίλων του Δάσους ε, Μπουσί κυρία Ντιμορτιέ εκπροσωπεί αυτήν την οργάνωση. Είμαστε δύο λοιπόν οργανώσει που έχουμε υποβάλει αυτήν την αναφορά και βρούμε κατόπιν αιτήματο των μελών των δύο αυτών οργανώσεων, συμπολιτών μα. Επίση, ε, είναι διαπερατό το υπέδαφο, δηλαδή είμαστε σε μια περιοχή, για να δούμε την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, είμαστε σε μια περιοχή που είναι ε, στο μετέχμιο ε, το, μιας περιοχής που είναι ε, ένα πέτρωμα με άργυλο και άμμο και πολύ μικρό πάχος έχει αυτή, αυτό το πέτρωμα και φτάνουμε στα 3 με 6 μέτρα εκεί από την ε, ε, από το χώρο ταφής, υπάρχουν ε, ρογμές αυτό το υπέδαφος, έχει καρστικό, είναι καριστικό το, το υπέδαφος στο σημείο αυτό και επομένως πάρα πολύ γρήγορα ε, μπορεί να διαφρωθεί. Αυτός λοιπόν ο καρστικός χαρακτήρας μας απασχολεί πάρα πολύ γιατί είμαστε πάνω από ουσιαστικά μία κοιλότητα που έχει βρεθεί εκεί. Γιατί λοιπόν ο νομάρχης του Λουαρέ έχει δεχθεί να γίνει εκεί αυτός ο Χίτα. Το 2009 ένας ε, εγκεκριμένος συντρογιολόγος κ. Μαζέ ε, έδωσε κάποια έγγραφα, έδωσε κάποια άλλα στοιχεία, προσαρτήματα, αλλά βλέπουμε σε αυτά τα έγγραφα ότι κάνει πολύ σοβαρά λάθη, δηλαδή δεν δέχεται ότι υπάρχουν κοιλότητες, ότι είναι καριστικό δηλαδή. Μιλά για ένα κενό 5 εκατοστών, αλλά εμείς έχουμε άλλα στοιχεία από μια τομή που έχουμε μας δείχνουν ότι υπάρχουν 10 και 50 εκατοστά. Άρα μιλάμε για κοιλότητα για μια, ένα σπηλώδη σχηματισμό. Και σε αυτή λοιπόν την περιοχή επίσης βλέπουμε ότι είναι 3 με 6 μέτρα κάτω από το χώρο αυτό, αυτή, αυτό το ειδικό πέτρωμα που σας είπα, το αργυλοαμόδες πέτρωμα. Άλλα λέει ο κύριος ε, ε, αυτός όμως το έγγραφό του. Επίσης βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και κανένα λατομείο ε, στο BC Σαν Lifar. Μόνο στο γειτονικό δήμο υπάρχει ένα τέτοιο λατομείο. Η μελέτη στην οποία λοιπόν στηρίχθηκαν και την οποία την έκαναμε σε πέντε μέρες ε, το 2009, στην οποία στηρίχθηκαν λοιπόν από την Ομαρχία, δεν γίνεται δεκτός ο σπηλαιώδη αυτός χαρακτήρα, δηλαδή ότι είναι καρστικό το υπέδαφος, ε, ούτε οι ε, χάρτες του BRGM και όλες οι άλλες ε, μελέτε που λένε ότι υπάρχει καρστικό υπέδαφος δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Βλέπετε τη γραμμή εκεί που δείχνει Επελέγει λοιπόν αυτό το τοπίο που υπάρχουν αυτές οι σπηλιές, υπάρχουν αυτές οι κοιλότητες που δεν έχουν όμως ε, ε, εξερευνηθεί. Βρέθηκαν 60 ε, εκατοστών κοιλότητες, μπορεί όμως πιο κοντά να είναι και μέτρο, ολόκληρα μέτρα αυτές οι, οι κοιλότητες, αυτές οι, οι σπηλιές. Και όταν γίνονται εργασίες εκεί βλέπουμε να υπάρχουν καθιζήσεις και αν είχε κατασκευαστεί και κάποιο οίκημα εκεί θα έπρεπε να είχαν ε, κλείσει οι κοιλώτες αυτές γιατί αλλιώς θα κατέρεε το οικοδόμημα. Αντίστοιχα λοιπόν, αν προσθέσει κανείς 25 ε, τόνους ε, τετραγωνικά μέτρα από πάνω, πάλι το ίδιο θα συμβεί, θα καθιζάνει το, το, το έδαφος αυτό. Και έχουμε και δύο μέτρα αυτό το αργυλώδε πέτρωμα, θα έχουμε όμως καθίσει, θα έχουμε κατάρρευση, και η εν λόγω τοποθεσία δεν είναι καθόλου καλά προσαρμοσμένη και δεν τηρεί και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Εδώ σας δίνουμε και κάποια έγγραφα μαζί με το είναι αναφορά μας για να σας δείξουμε πώς στο Λουαρέ όταν αυτή η καμπύλη, ο θόλος καταρρεύσει, τη σπηλιάς όλα τα από πάνω στοιχεία, 3 με 6 μέτρα πάχους, ε, θα πέσουν, θα διαραγεί, θα σχιστεί αυτή η μεμβράνη και έχετε ε, ένα παράδειγμα του φαινομένου που συμβαίνει συχνά όταν έχουμε κάποια κατασκευαστικά έργα, όπως έγινε για το, με το τραμ το 2011 στην Ορλεά ή και σε, μια, σε ένα παρεκκλήσι σε μεμά, πάλι κοντά σε αυτή την περιοχή. Εδώ βλέπετε το SC4, ε, αυτή την ε, γεώτρηση που είναι στην ανατολική γωνία του Χίτα και εκεί βρέθηκε αυτή η δεξαμενή για την διάλυση των ε, λιμάτων. Πρέπει να δούμε αυτή η σπηλιά τελικά, αυτή η κοιλότητα, πόσο μεγάλη είναι και αν υπάρξει σημαντική ή όχι κατάρρευση, καθίζηση. Έχουμε στείλει και άλλα στοιχεία πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως θα έπρεπε να σας δείξουμε τώρα κάποιες φωτογραφίες για να δείτε αυτό το χώρο, το φτωχύτα. Αυτό βλέπετε την ε, ε, μεγάλη ε, αυτή έκταση, τέσσερις ε, μονάδες καύσης, 80.000 ετών το χρόνο. Έχουμε και δύο χίτα 250.000. Εδώ βλέπετε το BCS Lifar, το συγκεκριμένο χίτα, αλλά με βάση ε, το σχέδιο για την ε, επεξεργασία αποβλήτων στο Λουαρέ είναι 110 με 120.000. Άρα έρχονται και από αλλού ε, τα, τα απορρίμματα για να φούν εκεί και αυτό είναι αντίθετο και με την οδηγία, την Ευρωπαϊκή Οδηγία. και στα βόρεια του δάσου της Σολιάνη βλέπουμε ότι τα απορρίμματα μιας πόλης που είναι από 160 χιλιόμετρα απόσταση έρχονται στις, στις ε, έρχονται στην, ε, στο χίτα του BC και υπάρχουν και ε, κάποιες άλλες τοποθεσίες που δεν, δεν τις εκμεταλλεύονται για την εξεργασία των αποβλήτων. Επίσης, αυτό τον χίτα που τον βλέπετε σε κάποιες φωτογραφίες, βλέπετε ότι εκεί προσελκύονται και πτηνά. Υπάρχουν δύο απόβλητα που πρόκειται από σούπερ μάρκετ, από την, διατροφική βιομηχανία, από τα ε, εστιατόρια και βλέπουμε ότι προσελκύουν τα πτηνά. Όμως η Ευρωπαϊκή Οδηγία το 99 στο άρθρο 5 λέει ότι θα πρέπει τα βιοαπόβλητα να αντιμετωπίζονται διαφορετικά, να ανακυκλώνονται, να επαναχρησιμοποιούνται με κάποιο τρόπο. Επομένως, ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει η ανάκτηση των δύο βιοαπορριμμάτων να επιταχυνθεί. Υπάρχουν και κίνδυνοι πυρκαγιάς, το αναφέρουμε και αυτό, για να σας πούμε ότι ήδη είχαμε πυρκαγιές επιτόπου Ε, δεν είναι ένα βέβαια θέμα το οποίο απαιτεί τις οδηγίες αυτής. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας λοιπόν το υπέδαφος, αλλά θα πρέπει να γίνουν και άλλες γεωτρήσεις από τον ε, νομάρχη. Θα πρέπει να ληφθούν και να συναχθούν τα συμπεράσματα και σίγουρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μην επεκταθεί αυτή η τοποθεσία. Τρία χρόνια ήδη έχει ξεκινήσει η μετάλλευση και αναμένεται να διαρκήσει 12. Ε, υπήρξε μια θετική γνωμοδότηση με 13 επιφυλάξεις ε, από τον ερευνητή, μια από τις οποίες λέω ότι δεν θα πρέπει στο μέλλον να επεκταθεί ο χώρος αυτός. Άρα δεν θα έπρεπε καν να έχει γίνει και αυτός ο Χίτα ή σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστούμε ε, που ε, δεχτήκατε την αναφορά και ελπίζω και εσείς να επιμείνετε μαζί μας ε, στο Γαλλικό κράτος και στο Ομάρχη ώστε να διορθωθεί η κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ζαμπρίσκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you very much. Ευχαριστώ τα προβλήματα των ε, αναφορών που αναφέρονται γενικώ ε, στα απόβλητα ε, είναι τα πλέον συνηθισμένα και συνήθως ε, δυσανασχετεί η περιοχή ε, και υπάρχει νομοθεσία η οποία είναι αρκετά ανοιχτή σχετικώς με αυτές. Γενικώ όμως μπορούμε να πούμε ότι η υγειονομική ταφή μπορεί μόνο να γίνει εάν βρίσκεται σε ένα σημείο με διορθωτικά μέτρα και δεν ε, δημιουργεί ε, σημαντικό περιβαλλοντολογικό κίνδυνο. Η απόφαση λαμβάνεται με ε, εξουσιοδότηση των κρατών μελών που δεν δίνει την άδεια εάν δεν βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ο αναφέρον μας δίνει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους ε, υποτιθέμενους κινδύνους αλλά η αρμόδια εθνική αρχή εξέτασε την περίπτωση και δύο φορές το θέμα κατέληξε στα δικαστήρια και στις δύο φορές απερίφθη και την πρώτη φορά και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον <clears throat> δεν έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει λεπτομερώς τους υποτιθέμενους κινδύνους για την υγειονομική ταφή οι οποίοι μας υποβάλλονται, ούτε ε, ούτε μπορεί να θεωρήσει ότι οι δικαστικές αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων παραβιάζουν την, ε, νομική, την ε, κοινοτική νομοθεσία. Οπότε δεν βλέπουμε κανένα λόγο να παρέμβουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος Μπουλό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον αναφέροντα για την ερώτησή του και για τη φροντίδα του του περιβάλλοντος. Όντως αυτός ο φάκελος παρουσιάζει ορισμένα ερωτηματικά τα οποία μπορούν να απευθύνονται είτε στην Επιτροπή είτε στον αναφέροντα. του, ε, η, ε, η σχετική ε, οδηγία έχει εφαρμοστεί και έχει τη 1999-31 και ε, έχει αξιολογηθεί επίσης όσον αφορά τα 25 μέτρα δηλαδή η πίεση στο υπέδαφο στην οποία είπατε ότι ε, εξασκείται είναι ένα λογικό ύψος και η Επιτροπή μπορεί να μειώσει αυτό το ύψος κατά τρόπον ώστε εάν και εφόσον μπορέσει να παρέμβει στην περίπτωση για να μην υπάρχει κατολίσθηση. Επίσης όσον αφορά την εκμετάλλευση για μία δωδεκαετία. Το ερώτημα είναι αν μετά τα 12 χρόνια ο βασικός ο κίνδυνος κατολίσθησης ε, και καφίζησης ε, που υπάρχει και ρηπάνσεως ε, των, υδάτων, των υπογείων υδάτων έχει συνυπολογιστεί. Και τέλος θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε ε, αξιολογήσει ε, την ε, κατάσταση των υδάτων στο Λουαρέ και αν η Γαλλία έχει εφαρμόσει το σεβασμό της, του περιορισμού της μετακινήσεως των αποβλήτων και ε, του θέματος των κατολιστήσεων και καθιζήσεων κατά τρόπον ώστε να μην υπάρξει λαπτική ενέργεια στα υπόγεια ίδια ε, διότι όπως είπατε προηγουμένως ε, καταλήγουν με αυτόν τον τρόπο εκεί πάρα πολλά απόβλητα τα οποία προέρχονται και από άλλους τομείς και όχι μόνο αυτά. Η κυρία Όκεν έχει στήσει πίσω το λόγο. Ναι, θέλω να προσθέσω κάτι όσα ακούσαμε πριν. Για μια ακόμη φορά εδώ έχουμε να κάνουμε με την οδηγία για τα λύματα και τα απόλυτα που δεν εφαρμόζεται. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν εδώ με ένα χώρο υγειονομικής ταφή αποβλήτων. Δεν ξέρω αν δεν κατάλαβα πολύ καλά. Πολύ κοντά όμως λέτε υπάρχουν εκεί υπόγεια ύδατα. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο να έχει πει η Επιτροπή Ευρωπαϊκή. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν μας αφορά ακριβώς. Γιατί έχουμε, ξέρετε, οδηγία, έχουμε νομοθεσία για τα απόβλητα. Είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτή η οδηγία. Και θα πρέπει να κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Πού υπάρχουν άλλες αναλλακτικέ λύσεις που να σέβονται αυτή την οδηγία. Διαλογή, αποβλήτων, ανακύκλωση, παναχρησιμοποίηση, όλα αυτά θα μπορούσε να ξαναχρησιμοποιηθεί, να ανακυκλωθεί αυτού του είδους, αυτού του από τα απόβλητα, τα απορρίμματα. Λέτε θα κάνουμε άλλη μία διαφορετική, σε μια διαφορετική τοποθεσία. Είπατε ε, χώροι δημιουργής ταφής, μα δεν, δεν ξέρω, και αυτά 25 μέτρα ο πρόεδρο ναι, πράγματι, δεν είναι μόνο αυτό που είπατε πολύ σωστά. Δεν έχουμε μόνο τι οδηγίε, έχουμε και την έκθεση. Ήμουν και εισηγητή. Θα θυμάστε, κύριε Άουκεν. Φαντάζομαι θυμάται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την έκθεση. Υπάρχει κάποιο άλλο συνάδελφο πριν δώσει το λόγο σε αναφέροντε. Μήπω θέλετε να απαντήσετε στα ερωτήματα όσων ε, έλαβαν το λόγο πρόσωπο της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ στα παραδείγματα ή μάλλον στα συμπληρωματικά σχεδιχεία που μπορώ να σας δώσω ότι όντως το Λουαρέ δεν ήταν καν γνωστό ότι υπάρχουν ε, βιολογικά απόβλητα ε, εις ε, την περιοχή αυτή και όταν συναντήσαμε τον νομάρχη εξεπλάγει για την άδεια αυτή που είχε δοθεί από τις υπηρεσίες τους ίσως δεν ήθελε να μην τη στηρίξει αλλά δεν ήξερε ότι ερχόντουσαν ε, και απόβλητα από άλλες περιοχές και όντως αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι δεν γνωρίζουμε παρόλο που έχω δουλέψει στην περιοχή ε, καμία υγειονομική ταφή στη Γαλλία που να είναι με ένα μόνο στοιχείο 25 μέτρα ύψος και πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρό και υπάρχουν πολλές ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο έγινε αποδεκτή ο φάκελος που υπέβαλε ο αναφέρον διότι ε, ενδεχομένω εάν καταρρεύσει όλο αυτός ο όγκος θα, μπορέσει, θα σπάσουν οι μεμβράνες και ε, θα ρηπανθούν ε, τα υπόγεια ύδατα και θα καταλήξει το πρόβλημα και στον ποταμό Λίγυρα. Αλλά εφόσον απευθυνόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το πράξαμε διότι δεν ε, καταλαβαίναμε για ποιο λόγο τα διοικητικά δικαστήρια στη Γαλλία δεν είχαν ε, δεχθεί αυτόν τον επικίνδυνο χαρακτήρα. Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την ε, ε, αυτό το θέμα, αν συμφωνείτε, για επιπλέον ε, πληροφορίες και για να αξιοποιήσει κανείς ε, ορισμένα στοιχεία και για να έχουμε και περισσότερες απαντήσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Μάργαρετ έχει το λόγο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε για τα υπόγεια ύδατα απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ακούσουμε και τι έκαναν για να κοινοποιήσουν ότι υπάρχει οδηγία και ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάποια καινοτόμα μέτρα για να αλλάξει όλη η στρατηγική που ακολουθείται με τη χρήση χήτα. Κάψης θα ήταν ακόμα πιο ανοητή η λύση. Αλλά είναι ένα κομμάτι του να συμμορφωθούν με τις οδηγίες. Εάν θα μπορούσαμε λοιπόν πάνω σε αυτό να το, να το διαφωτίσει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε μια απάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει στην κυρία Όκεν ή μπορούμε να περιμένουμε πληροφορίε που θα μα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Σαφέ ότι θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Δεν ξέρω αν οι, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουν να πούνε κάτι. Αξιότιμα μέλη από αυτά που ακούω, είδα ότι διάφορες απόψεις εκφράστηκαν. Οι ερωτήσεις αποκλίνουν από την αναφορά. Η αναφορά αφορούσε την τοποθεσία της χωματερής. Από αξιότιμα μέλη άκουσα ότι τίθεται θέμα της όλης διοργανώσεως διαχειρήσεις αποβλήτων τουλάχιστον στη Γαλλία ή τουλάχιστον αυτή την περιοχή της Γαλλίας. Μπορούμε να δώσουμε και άλλες πληροφορίες αλλά σε αυτή τη φάση μπορώ να πω ότι τα κράτη-μέλη έχουν μεγάλη ελευθερία σχετικά με αυτό. Πρέπει να περιορίσουν τη χρήση χωματερών για βιοδιασπόμενα απόβλητα. Θα πρέπει στο μέλλον να συμμορφωθούμε στόχους για ανακυκλώσιμα απόβλητα, αλλά είναι στόχοι που τίθενται σε επίπεδο χώρας Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ. Ορίστε. Η κυρία Όκεν. Πολύ δημιουργική ερμηνεία της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκπλήσωμε λίγο, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι τώρα. Τι κάνουν όμως για να εφαρμοστεί η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην λένε είναι εθνικό στόχο μέχρι να βρεθεί λύση για τα πάντα και μετά να πούν κάτι άλλο. Δεν θέλω απάντηση τώρα. Δεν θέλω να ακούσω κι άλλη δημιουργική εντό εγωγικών απάντηση. Εφάνταστη απάντηση. Θέλω να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει κάνει για να ξεκαθαρίσει στους εκπροσώπους της περιοχής πρώτα και της χώρας μετά ε, τι πρέπει να κάνουν να με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μου φαίνεται πολύ καλό και καλά κάνεις και ζητάς αυτές τις πληροφορίες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή και βέβαια να ζητήσουμε από την Ομορφία πληροφορίες σε σχέση με αυτά που ακούσαμε σήμερα. Και μετά θα μας απαντήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία, περνάμε λοιπόν στην τροπολογία, στην αναφορά η 7 έχει ακυρωθεί. Έχουμε λοιπόν αναφορές για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπαρθμόν 8 στην ημερήσια διάταξη. Είναι η αναφορά από Ντανιέλ Μαριάν Γιώργα, Ρουμανική Ιθαγένεια, για τα εικαζόμενη παραβίαση του Ισπανικού Συντάγματο σε σχέση με τι υποθήκε που συστήνονται για την αγορά ακινήτων. Έχουμε επίση την αναφορά 179 του Χωσέ Μανουέλ Άλβαρεθ Μαρτίν, Ισπανική Ιθαγένεια, για την καθιέρωση και αποδοχή Τη έννοια datio in solutum, μεταβέσα αντιπληρωμή στην Ισπανία σε περιπτώσει εξώσεων. Και τρίτη αναφορά, η υπαριθμών 644 από το Χωσέ Μανουήλ Μαρτίν Άλβαρη. Ισπανική θα γίνει και αυτό σχετικά με τι πρακτικέ συνυπόθηκων δανείων και την καθιέρωση τη έννοια τη μεταβίβαση αντιπληρωμή datio in solutum στην Ισπανία. Ποιο θα λάβει το λόγο? Ποιος θα λάβει το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? ο κ. και κάπως έτσι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτές οι τρεις αναφορές ομαδοποιήθηκαν. Διαταφορούν λίγο πολύ το ίδιο ζήτημα. Οι τρεις αναφέροντες, ή πλέον επακριβώς δύο αναφέροντες, διότι μία, δύο αναφορές απεστάσαν τον ίδιο άνθρωπο. Αφορούν λοιπόν το πρόβλημα διαδικασιών ε, κατασχέσεων στην ε, Ισπανία και πιο συγκεκριμένα αναφέρονται διότι επιτρέπει αυτές τις διαδικασίες η Ισπανική κυβέρνηση σαν αποτέλεσμα μίας αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων από τους καταναλωτές. Ζητούν οι αναφέροντες η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει και να πιέσουν τη Ισπανική κυβέρνηση εισάγει το datio isolusum, δηλαδή τη διαδικασία διαπληρωμής ε, στον Ισπανικό νόμο. Ε, αναλύσαμε λεπτομερώς τις αναφορές και συμπεράναμε ότι δεν εμπίπτει της της Ευρωπαϊκής Ενώσης αυτό. Οι διαδικασίες κατάσχεσης αντιμετωπίζονται εθνικής βάσεως, ρυθμίζονται εθνικά. Το ίδιο και για τον Τάτιον Σολούτον. Για τη λύση αυτή. Τούτου λεχθέντος παραδέχομαι ότι εξετάζουμε προσεκτικά το όλο πρόβλημα προετοιμαζόμενοι για την οδηγία για πιστώσει αστεγαστικά δάνεια. Ετοιμάσαμε ένα έγγραφο ο αναλύει τα μέτρα που μπορούν να σταματήσουν να εμποδίσουν διαδικασίε κατάσχεση στα κράτη-μέλη. Ήταν ενημερωτικό όμω το έγγραφο. Παρουσίαζε τι πρακτικέ που ακολουθούνται στα κράτη-μέλη. Ένα είδο προσανατολισμού, αν θέλετε, για τι δημόσιε διοικήσει ήταν. Όπω προανέφερα, σε κάποιο βαθμό για να αποφευθεί αυτό το πρόβλημα στο μέλλον, όπως τα γνωρίζετε, προτείναμε την οδηγία για τις ε, πιστώσεις για στεγαστικά δάνεια που συζητιέται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αλλά εν λόγω οδηγία αφορά όμως την προ-συμβασιακή φάση και δεν παρεμβαίνει στην συμβασιακή φάση. Δηλαδή μεταξύ ε, του πιστωτού και του δανειολήπτου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα, δεν μπορεί να παρέμβει στο συγκεκριμένο τομέα. Ευχαριστώ κύριο Μέγερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, λυπούμε που δεν παρίστανται οι αναφέροντες. Είναι ένα ζήτημα που πραγματικά δημιουργεί ένα πολύ έντονο κοινωνικό πρόβλημα στην Ισπανία. Η κρίση πλήττει πάρα πολύ βαριά και την Ισπανία και όχι βέβαια κάποια άλλα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ερωτήσεις προς την... και έχω και εγώ υποβάλλει. υποβάλει, μου απάντησαν εγγράφος από την Κομισιόν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να ληφθούν νομοθετικά μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκεί όταν δηλαδή έθεσα τα ερωτήματα μου απάντησαν αυτό. Εγώ όμως νομίζω ότι καλό θα ήταν να πρέπει να εναρμονίσουμε, να ρυθμίσουμε αυτή την έννοια «datium solutum» μεταβίβαση αντί και να έχουμε έτσι μια γενική προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποια κράτη που έχουν ρυθμίσει, όπως Πορτογαλία, Γερμανία, ε, Γαλλία. Εγώ θα έλεγα να καλέσουμε τους αναφέροντες. Έχουμε 517 εξώσεις ε, στην Ισπανία και όταν βλέπουμε να χάνουν την δουλειά τους ε, οι άνθρωποι και να έχουν ένα στεγαστικό δάνειο που δεν μπορούν να το πληρώσουν, ε, τους διώχνουν το σπίτι τους, ε, τους κάνουν έξωση. Και παρόλα αυτά όμως πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν και το στεγαστικό δάνειο σε αντίθεση με τα κράτη που σας ανέφερα που έχουν ρυθμίσει με αυτήν την αρχή ντάτη σε όλο το θέμα. Έγινε μια πρόταση για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε την κατάσταση. Υπήρξε μια πρόταση βασιλικού διατάγματος, αλλά επειδή στα χέρια των τραπεζών πλέον επαφίεται το να ρυθμίσουν αυτή τη ε, μεταβίβαση αντιπόλησης, ξέρουμε τι κάνουν οι τράπεζες. Στο δεύτερο εξάμεινο ε, την, ε, του, χρόνου είχαμε, το προηγούμενο, είχαμε 517 εξώσεις καθημερινά. Με αυτή την έννοια και επειδή έχουμε εμπειρίε, ξέρουμε, μάλιστα και πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναγνώρισε, είχαμε μια συζήτηση στην Επιτροπή μας, αναγνώρισε την ανάγκη να υπάρξει νομοθεσία για αυτό το κενό που υπάρχει παραδείγματο χάρη για τα βιβλία σε Και εδώ υπάρχει ανάγκη όχι μόνο για την Ισπανία αλλά και για άλλα κρατημέλη που δεν έχουν ρυθμίσει αυτή την αρκετά την Σολούτου. Πρέπει να γίνει αυτή η θετική προσπάθεια και νομίζω ότι πρέπει να καλέσουμε και τους αναφέροντες, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έρθουν εδώ στις Βρυξέλλες και να έχουν μια συζήτηση ώστε πραγματικά να υπάρξει πρόοδο και να έχουμε την νομοθεσία που θα ρυθμίσει με ομοιογενή τρόπο και σε όλα τα κράτη-μέλη την αρχή ντάτιο Είχαμε αυτό το παράδειγμα πρόσφατα δηλαδή σε σχέση με την υποχρέωση της δημοσίευσης των βιβλίων σε μπράι. Υπήρξαν κάποια ελάχιστα κριτήρια που δεν υπήρχαν. Έγινε αυτή η συζήτηση. Καταφέρουμε να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Αφού το κάνουμε αυτό το θέμα, καλό θα ήταν να το κάνουμε και στην προκειμένη περίπτωση. Απλά λέω κύριε Πρόεδρε να παραμείνει ανοιχτό το θέμα, να καλέσουμε τους αναφέροντες. Ουσιαστικά γι' αυτό το λόγο να μείνει ανοιχτή αναφορά. και όπως ζητούν και αναφέρονται να ξεκινήσει όλη η συζήτηση για το πώς θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε το ζήτημα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος, τρία πράγματα θέλω να σας πω κύριε Μέγια. Πρώτα απ' όλα ότι οι αναφέροντες από το Μιλένη Γραμματεία έχουν ενημερωθεί, ε, ενημερώθηκαν εγκαίρως. Όχι λέτε και δεν μπορούσαν. Τέλος πάντων, εσείς μου λέτε όχι. Ε, θα το δούμε. Μπορούμε στους συντονιστές να το συζητήσουμε. Η γραμματεία μου λέει ναι, εσείς λέτε. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα τους δώσουμε πάντως τη δυνατότητα γιατί όπως ξέρετε οι κανόνες λένε ότι εάν ένας βουλευτής θέλει να μείνει αναφορά ανοιχτή, μένει ανοιχτή. Παρά το ότι όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ακούσατε κι εσείς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Υπάρχει το άρθρο 18 που λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να ρυθμίζουν την ε, μεταβέση αντιπόλησης και μας πενθυμίσατε κι εσείς ότι ε, το Υπουργικό Συμβούλιο της 9 η Μαρτίου ενέκρινε αυτό το βασιλικό διάταγμα για την ε, μεταβέση αντιπόλησης, μετά υπήρξαν ερμηνείες, εσείς κτλ. Πάντως το των λεχθέντων θα έχουν τη δυνατότητα αναφέροντας να μας τα πούν από κοντά Μπορείτε να συστήσετε πάντως με την γραμματή για να ξεδιαλύνουμε γιατί ε, δεν ήρθαν οι αναφέρτες. Ε, δεν ξέρω ποιος ε, έχει τις πιο επίκαιρες πληροφορίες, εσείς η γραμματεία, τέλο πάντων μπορείτε να το δείτε διμερώς. Τούτου λεχθέντο, περνάμε στην επόμενη αναφορά, νέα στην ημερήσια διάταξη, αναφορά από τον Τζον Πάρσο Βρετανική Ιθαγένειας, εξονόματος τη Costa del Sol Action Group, σχετικά με την έλλειψη διαδικασιών υποβολή καταγγελιών και υπηρεσιών διαμεσολάβηση στο χρηματοοικονομικό τομέα στην Ισπανία. Παρακαλώ, πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Ε, Πρόεδρε, αναφέρει ο αναφέρον τι έγινε με κάποιους επενδυτές στην Νότια Ισπανία. Έλαβαν διάφορες σηματοσυντικές υπηρεσίες από συμβούλους ε, το 2001. Αναφέρονται εμπειρίε όσον αφορά του παρόχου υπηρεσιών και όσον αφορά τι χρηματοσυντικές υπηρεσίε οι περισσότεροι ήταν σύμβουλοι που δεν ρυθμιζόταν και δεν ήταν καταχωρημένοι και τα προϊόντα και υπηρεσίε σε πολλέ περιπτώσει, διάφορα αξιόγραφα και διάφορε επενδύσει, επενδυτικά προϊόντα αναφέρονται στην αναφορά. Στην αναφορά ο αναφέρον αναφέρει την έλλειψη διαδικασιών προσφυγής και διαμεσολαβητού στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να δώσει κάποιε πληροφορίε και παρατηρήσει από αυτού. Σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παραχή συμβουλών που δεν είναι οι αρμόζωσε από διάφορου συμβούλου που δεν ρυθμίζονται για διάφορα προϊόντα και την έλλειψη διαδικασιών ε, διαμαρτυρία, καταγγελία στην Ισπανία. Σχετικά με αυτό, θα ήθελε να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σχετικά με αυτό διάφορε νομοθετικέ πράξει και πρωτοβουλίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, θα μπορούσαν να ταιριάξουν. Η παροχή συμβουλών αυτών καλύπτει το μύθι, την οδηγία για τις αγορές και χρηματοπιστωτικά μέσα που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007 και πέρα. Οι επενδυτικέ εταιρείε και οι τράπεζε που δίνουν επενδυτικέ συμβουλέ πρέπει να συμμορφωθούν με διάφορου κανόνε όσον αφορά του πελάτε του. Κυρίω όσον αφορά ε, του πελάτε λιανικού εμπορίου, θα πρέπει να ενημερώνουν του πελάτε όσον αφορά τα διάφορα χρηματοστικά μέσα που προτείνονται και τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν. Επιπλέον, θα πρέπει να πάρουν τι πληροφορίε για τα χρηματοστικά μέσα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των πελατών, γνώση, εμπειρία, οικονομική του κατάσταση, στόχο, για να συστήνουν τα χρηματοστικά μέσα τα οποία είναι κατάλληλα για κάθε πελάτη. Τώρα τα κράτη-μέλη μπορούν να εξαιρέσουν κάποιε επενδυτικέ συμβουλέ από το πεδίο εφαρμογή του MIFID υπό τη στιγμή που ρυθμίζονται και ελέγχονται εθνικό επίπεδο. Όμω, καμία, κανένας δεντολογικός κώδικας δεν προβλέπεται από την οδηγία. Και τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται αλλά δεν υποχρεούνται σύμφωνα τη νομοθεσία να καθορίσει δικασίες για, διευθέτηση, για εξώδικες διευθετήσεις διαφορών. Λοιπόν, όσον αφορά την νομική κατάσταση που κρατεί και ενδεχόμενε παραβίαση των κανόνων περί επενδυτικών συμβουλών και κανόνων MIFID, ο αναφέρον θα πρέπει να στραφεί προ την αρμόδια αρχή, εποπτική αρχή της Ισπανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη συνθήκη έχει την εξουσία να παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το ένα κάτω μέλο υπό την προπόθεση ότι υπάρχει παράβαση όσον αφορά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού νόμου, αλλά που δεν έχει άμεση εξουσία να κινηθεί κατά εθνικών χρηματοστικών φορέων που δεν πληρούν τι υποχρεώσει όσον αφορά ε, ατομικέ υποθέσει, ξεχωριστού πελάτε. Σε αυτή την περίπτωση, ο αναφέρον ίσω θα ήθελε να εξετάσει τον κατάλογο των διαφόρων φορέων διαθέτηση διαφορών, ούτω ώστε να θεωρήσει κατά πόσο η υπόθεσή του μπορεί να αποτελέσει δικαίωμα προσφυγή κατά του αρμόδιου φορέα τη Ισπανία. Και θα δίναμε τη συμβουλή στον αναφέροντα να δει κατά πόσο εξωτερική νομική συμβουλή θα ήταν δεγμένη η λύση. Στην τωρινή κατάσταση υπάρχουν νομοθετικές πράξεις και πρωτοβουλίες που καλύπτουν συμβούλους που δεν είναι καταχωρημένοι και δεν ρυθμίζονται και δεν ελέγχονται για να μειωθούν αρνητικά αποτελέσματα όπως αυτό που αντιμετωπίζει ο αναφέρον. Το MIFID αναθεωρείται. σε νομοθετική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για βελτίωση των κανόνων για προστασία των επενδυτών και η αύξηση εμπιστοσύνη των επενδυτών και παροχή συμβουλών επενδυτικών αποφορής καλύπτονται τρόπο. Πρώτα, οι φορεί που αδειοδοτούνται σύμφωνα με το MIFID υπόκεινται σε περαιτέρω αδειοδότηση και απαιτήσει για δεντολογική συμπεριφορά επιχειρηματική. Δεύτερον, φορεί που εξαιρούνται από του κανόνε MIFID υποχρεούνται να συμμορφωθούν με ουσιαστικέ απαιτήσει, ανάλογε τουλάχιστον με αδειοδότηση και απαιτήσει δεντολογικέ. Τρίτον, παροχή υπηρεσιών χωρί αδειοδότηση ε, συνεπάγεται κυρώσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει επιπλέον πρόσφατη υιοθέτηση της πρότασης για βελτίωση διαφάνειας όσον αφορά τις επενδυτικές υπηρεσίες λιανικού εμπορίου και μετά υιοθέτησε πρόταση για οδηγία για συμφωνίες επενδυτικές όσον αφορά κατοικίες. Υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2011 εν λόγω πρόταση. Κλείνοντας, η αναφορά αναφέρεται στην παροχή ακαταλήλων συμβουλών από διαφόρους σύμβουλους, οι οποίοι δεν ελέγχονται και καλύπτουν διάφορα προϊόντα και έλλειψη δυνατοτήτων προσφυγής. Ξαναλέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί άμεσα να ασχοληθεί με το θέμα, δεν έχει τέτοια εξουσία όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζουν οι Ισπανικές αρχές το πρόβλημα του αναφέροντος και τους πελάτες του τομέα της λιανικής, όμως διάφορες νομοθετικές πράξεις και πρωτοβουλίες όπως προανέφερα καλύπτουν την παροχή χρηματοδοτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλε αυτέ οι πρόσφατε πρωτοβουλίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ανέβησαν πρόσφατα θα ισχυροποιήσουν την προστασία των επενδυτών και των πελατών παρεχόντων χρηματοστικών υπηρεσιών για να αυξηθούν οι κυρώσει την παραβίαση των νόμων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και θα ενηθούν τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν εξώδικες διαδικασίες για τη διευθέτηση των διαφορών και καταγγελιών. Ευχαριστώ. Θέλει το λόγο παρακαλώ και συνάδελφο για αυτό το θέμα. Όχι. Άρα, αν κανείς δεν θέλει το λόγο, σημειώνουμε τις ε, εξηγήσεις της Κομισιόν και αφήνουμε το θέμα ως έχει. Θα μπορούσαμε ίσως να ενημερώσουμε την Επιτροπή, την Επιτροπή Εσωτερικού Εμπορίου, ΙΜΚΟ, για να το εξετάσουν κι αυτοί. Υπάρχει αντίρρηση. Όχι. Ωραία. Έτσι λοιπόν θα γίνει. Ολοκληρώσαμε τα σημεία της ημερησίας διάταξης για σήμερα. Πέντε ξεκινάει η συνέντευξη των δοστών. Μπορούμε λίγο να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα ή να περιμένουμε για να εντοπίσουμε αυτούς που λείπουν. Ποιοι λείπουν. Όχι. Πέντε η ώρα, μου λέει ο γραμματέα. Ναι, λέει κυρία, και αλλιώ θα μείνετε εσεί και εγώ και θα τα αποφασίσουμε οι δυο μα όλα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, λέει ο πρόεδρο, αλλά ίσω. Καλό θα ήταν να περιμένουμε τους άλλους συντονιστές. Πέντε λοιπόν, πέντε η ώρα θα συνεχίσουμε.